σιδηροδρομικά δίκτυα και δημόσιε υπηρεσίε στις μακροπεριφέρειες του Δούναβη και της Κρέτσου. Ο λόγος στην Επιτροπό Κορίνα Κρετσού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που έχετε προβλέψει το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. ο ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών στη βελτίωση παροχή συνδρομικών υπηρεσιών στις μακροπεριφέρειες του Δούναβη και τη Αδριατικής είναι αυτό που θα μας αποσχολήσει. Την περασμένη εβδομάδα έλαβα μέρος στη συζήτηση για την ε, μακροπεριφέρεια των Άλπαιων στον Μπούντο της ε, Σλοβενίας. Είναι η τέταρτη φορά που συζητάμε για μια, για μια στρατηγική μακροπεριφέρειας και μας δείχνει αυτό το παράδειγμα ότι οι μακροπεριφερειές είναι πολύ σημαντικές για την κατάρτιση σωστών στρατηγικών. Μπορούμε με τον τρόπο αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα διάφορα προβλήματα, βλέποντας την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή. Αυτού του είδους η συνεργασία είναι πολύ σκόπιμη για την πρόοδο των διάφορων περιφερειών και στη συγκεκριμένη περίπτωση με την ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων. Οι στρατηγικές του Δούναβη και της Αδριατικής έχουν εντοπίσει τις υδροδρομικές υπηρεσίες ως προτεραιότητα. Υπάρχουν κενά, τεράστια κενά ε, και διαφορές μεταξύ, της παροχής, μεταξύ των διάφορων περιοχών στην παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών και ως προς το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης. Τα παλιά κρατημέλη, ε, Ιταλία, Γερμανία και Αυστρία, έχουν πολύ καλύτερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Ενώ υπάρχει περιθώριο βελτίωση ενώ στα κράτη-μέλη, όπω η Δημοκρατία τη Τσεχία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, η κατάσταση δεν είναι το ίδιο ικανοποιητική. Όμω είναι καθοδόν προ μια περαιτέρω βελτίωση. Τώρα για τι χώρε εκτό Ευρωπαϊκής Ένωση, οι συντηροδρομικέ υπηρεσίε έχουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και επενδύσει. Σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πλέον η ώρα να ληθούν μέτρα για να στηριχθούν οι συνδυοτρομικές υπηρεσίες και γενικότερα οι δημόσιες υπηρεσίες της περιφέρειας αυτές. Θα πρέπει να στοχεύσουμε συγκεκριμένες πτυχές. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ισχυρή και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να πετύχουμε τις στρατηγικές ε, στις μακροπεριφέρειες. Έπειτα πρέπει οι χώρες να συνεργαστούν στενά για να ε, υλοποιήσουν τις υδροδρομικές μεταρρυθμίσεις, όπως την αποσύνδεση των ε, υποδομών και την θέσπιση κανόνων. Επίσης, πρέπει να επενδύσουμε σε προγράμματα αποκατάστασης και αναβάθμισης για τις υδροδρομικές συνδέσεις και τα διάφορα σημεία που λείπουν στην αλυσίδα ως προς τον συντονισμό για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκτιμόμενη αξία του δικτύου TNT είναι ακριβώ και το τέλειο πλαίσιο για τέτοιου είδου επενδύσει. Από την άλλη, όμω, κυρίε και κύριοι μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, γνωρίζουμε όλοι ότι η συνεργασία μεταρρυθμίσει και επενδύσει στου υδροδρόμου δεν επαρκούν. Δεν μπορούμε μόνο με αυτό το, με αυτή τη στρατηγική να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Πρέπει να προβλέψουμε και επενδυτικά προγράμματα καθώς και σωστέ δομές διακυβέρνηση, αλλά και διασυνοριακές διαδικασίες να απλοποιηθούν. Πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταλήξουν σε συμφωνία σε ό,τι αφορά την εξή σημαντική αρχή. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι συμβάσεις τους στον τομέα των σιδηροδρόμων θα βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν πολλές σοβαρές προκλήσεις σε αυτόν τον χώρο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πόροι που διαθέτουμε ε, χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Πριν από τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση, την τέταρτη δεσμή μέτρων για του σιδηροδρόμου και πιστεύουμε ακλόνητα ότι ω συνομοθέτε εσεί και εμεί μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την πρόταση αυτή. Ε, Όπω προείπα, έχουμε ήδη πετύχει πολλά στις μακροπεριφερειακές μας στρατηγικές, οπότε είναι τώρα πλέον η στιγμή αυτές οι αρχές να, να πάρουν σάρκα και οστά με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες κινήσεις για να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών. Δηλαδή, καλύτερε δημόσιες ιδεροδρομικές υπηρεσίες, πιο αποτελεσματικές. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τι ε, σα. Uh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Οι μακροπεριφερειές είναι μια θετική πρωτοβουλία γιατί οδηγούν σε καλύτερο συντονισμό και συνοχή των διαφόρων περιφερειών που ανήκουν σε μια μακροπεριφέρεια. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα λεφτά να μην ε, φτάσουν εκεί πέρα παρά μόνο ελάχιστο ποσοστό. Αλλιώ θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Χρειάζεται συντονισμός σε επίπεδο Κομισιών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμφωνήσουν ε, να διοχετεύσουν τα λεφτά σε έργα συνεκτικά που θα γίνουν σε πολλές χώρες μαζί. Όσον αφορά τον Δούναβη και τα Βαλκάνια, η πρωτοβουλία της Κομισιόν να επεκταθεί το δίκτυο των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφόρων στα Βαλκάνια είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό για να δημιουργήσουμε διαδρόμους με έργα που θα τα βάζουν όλα αυτά στην θέση που πρέπει στην Κωνσταντζα, στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και με τα ελληνικά λιμάνια γιατί τελικά τα εθνικά σχέδια καταλήγουν σε διαδρόμους. Και έχουμε λοιπόν την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού πακέτου και επίσης πρέπει να επαναφέρουμε τα κονδύλια της Εύση στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ η κυρία Τσαπαρτέλη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κρέτσου, χαίρομαι που γίνεται αυτή η πολύ σημαντική συζήτηση για τη Ρουμανία και την Ανατολική Ευρώπη. Η Ρουμανία και η Αυστρία ήταν οι πρώτες ε, χώρες ε, που συνέδεσαν ε, τους σιδηροδρόμους τους και ζήτησαν από την Κομισιό να αναπτύξει μια στρατηγική για τον Δούναβη. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη για κινητικότητα, για αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, ε, την ποιότητα του νερού και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχουν κοινέ προκλήσεις βεβαίως, αλλά η οικονομική ανάπτυξη διαφέρει, οπότε χρειαζόμαστε εργαλεία για περισσότερη κοινωνική συνοχή και εδαφική συνοχή το master plan της Ρωμανίας είναι ένα τέτοιο εργαλείο. και βεβαίω ε, πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες επενδύσεις στις υποδομές. Το master plan αυτό υιοθετήθηκε από τη ρουμανική κυβέρνηση και μετά εγκρίθηκε από την Κομισιόν μετά από διαπραγματεύσεις. Ε, τα έργα υποδομών αυτά είναι προτεραιότητες ε, που ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες της Ένωσης για έναν ενιαίο χώρο μεταφορών. Γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω πως αυτή η συνοχή μεταξύ περιφερειακής πολιτικής και μεταφορικής πολιτικής υπάρχει στην περιοχή του Δούναβη. Και έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εδαφική και κοινωνική συνοχή και να κλείσουμε κάποια κενά που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία να έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πράγματι ε, έχουμε ως βασική ελευθερία την ελεύθερη διακίνηση ε, προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Και βεβαίως ε, ε, προσπαθούμε να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη με το σιδηροδρόμο αλλά δεν είναι δυνατόν ακόμα γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις μακροπεριφέρειες είπατε πως είναι προτεραιότητα η σιδηροδρομική σύνδεση ε, και ε, βέβαια εδώ πέρα λείπουν πάρα πολλά πράγματα δεν μπορούμε να ενώσουμε όλα τα νησιά καλό θα ήταν για τα νησιά της Αδριατικής αλλά δεν μπορούμε Έχουμε λοιπόν ελλείψεις. Η μακροπολιτική λοιπόν έχει στόχο να ενώσει ό,τι μπορεί. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα χάρτη που έχουμε αναπτύξει για διαδρόμους σε ολόκληρη την Ευρώπη για τις διασυνδέσεις. Θα επικεντρωθώ σε τρεις διαδρόμους που είναι σε αυτή την περιοχή. Ο ένας είναι ο διάδρομος ε, Αδριατικής ε, Βαλτικής ε, με 16 διελεύσεις ε, συνόρων. Έχουμε πάρα πολλές στενοπούς, κυρίως στην Πολωνία και στη Σλοβενία. Εκεί πέρα δεν μετακινεί ο κόσμος εμπορεύματα με τον σιδηρόδρομο και απαιτούνται λοιπόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις που δεν μπορεί κανείς να πληρώσει και βλέπουμε πως αν θέλει να πει κανείς από την Αθήνα μέχρι το Αμβούργο πρέπει να περάσει έξι φορές από υδατοφράξη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και στον Δούναβη μέχρι τον Ρήνο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα επίσης και εμπόδια. Και στην Ρουμανία υπάρχει σοβαρή ανάγκη εξυγχρονισμού. Και θεωρώ πως θα πρέπει να επιτύχουμε βελτιώσεις στην πολιτική για τις ε, ε, μακροπεριφέρειες. Σας ευχαριστώ. Κρέμερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πριν από λίγου μήνε είχαμε τη διάσκεψη στο Παρίσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε πως ε, ανέλαβε κάποιες δεσμεύσεις, οποίε πρέπει τώρα να τι εφαρμόσουμε. Η κυκλοφορία ε, είναι υπεύθυνη για το 25% των εκπομπών και είναι ο μόνος κλάδος όπου έχει αυξηθεί οι συγκοινωνίες. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει η κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι θέμα που αφορά το μέλλον, γι' αυτό πρέπει να συνδεθούν και οι περιφέρειες, ε, οι περιφερειακές. Και μην κάνετε πάλι το λάθος της ε, Πορτογαλίας. Πριν από 10 χρόνια σταμάτησαν, έκοψαν σιδηροδρομικές γραμμές ε, γιατί θα πήγαιναν όλοι με τα μάξι, τώρα δεν έχουν λεφτά για τα μάξι και η κινητικότητα έχει καταστραφεί. Κοιτάξτε, Λέτε εδώ πέρα πω 30 με 40% των στερεοδρομικών γραμμών στη Ρουμανία πρέπει να κλείσει. Αποφάσισε η κυβέρνηση και συμφωνεί η Κομισιόν. Έτσι δεν θα επιτύχετε ποτέ τους κλιματικούς στόχους. Οπότε προτεραιότητα πρέπει να έχει ο σιδηρόδρομο. 60% των διαρθρωτικών ταμείων πάνε στους δρόμους και 20% πηγαίνουν στους Πρέπει να αλλάξει αυτό, όχι να κλείνεται σιδηροδρομικές γραμμές. Και βεβαίως και οι μικρές διαδρομές παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί 90% των επιβατών ταξιδεύουν λιγότερα από 50 χιλιόμετρα. Μην σκέφτεσαι μόνο τα μεγάλα έργα, όχι μόνο τα διευρωπαϊκά. Οι διασυνδέσεις να γίνουν ένα δίκτυο. Αυτό πρέπει να γίνει. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Σιδηρόδρομο, ε, είναι μια κουρελού και οι τρύπε είναι ακριβώς στα σύνορα πρέπει ακριβώς να υπάρξουν αυτές οι διασυνοριακές συνδέσεις που καταστράφηκαν στη μεταπολεμική εποχή, στον πόλεμο δηλαδή και δεν φτιάχτηκαν. Δεν είναι δυνατόν να λέτε κλείνω 30 με 40% των σειροδρομικών γραμμών της Ρουμανίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κράμερ, Θυμάμαι ότι τον Ιούνι ε, κάναμε ήδη στην Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου μια αντίστοιχη συζήτηση. Θυμάστε τι είπε και ο εκπρόσωπος της Ρωμανικής Κυβέρνησης ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και από τη ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΤΡΑΝΕ μας είπε ότι δεν πρόκειται περί αυτού ότι θα πάυσουν να λειτουργούν 30 έως 50% των ε, διασυνδέσεων, ε, των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων. Θέλουν να επιδιώξουν την βελτιστοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών και επειδή εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα δίκτυα, είπα ότι στην Γαλλία παραδείγματο χάρη έχουν σταματήσει να λειτουργούν πολύ περισσότερες σιδηροδρομικές γραμμές από ότι στην στην ε, Ρουμανία. Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο και ενιαίο σειροδρομικό δίκτυο και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Ε, ε, σας παρακαλώ να μην παραπλανάτε με τις πληροφορίες που δίνετε. Έχω μάθει το ότι γίνεται, γνωρίζω ότι στη Ρουμανία γίνεται μεγάλη συζήτηση για το εάν η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης θα αναγνωριστεί από το Κοινοβούλιο ή όχι και στην Κομισιόν το συζητάνε. Και εγώ γνωρίζω πως στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουν κοπεί πολλές σιδηροδρομικές γραμμές και το πολέμησα και αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει η χώρα. Ο σιδηρόδρομος είναι το μέλλον και μόνο με το σιδηρόδρομο θα σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Τα παιδιά μας και τα παιδιά τους να έχουν προοπτική. Αν όμως λέμε τώρα ότι θέμε να γίνει καλύτερο το δίκτυο και μετά κόβουμε 30 με 40% των γραμμών, αυτό δεν είναι βελτίωση, είναι καταστροφή που πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ. μισή λεπτό, Τζιλ. Ευχαριστώ. Ε, ε, για να το πω με τα περίφημα λόγια του Μπίσπεν καλά, τα προσαρμόσω στην 21ο αιώνα, ε, όπως λένε οι γραφειοκράτες, δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτά τα δίκτυα για να έχουμε εδαφικές συνέργειες και να μειώσουμε τις εδαφικές και γεωγραφικές ανισότητες. Παγκοσμιοποίηση, δηλαδή σε μία άλλο ένα και μεγαλύτερη και στενότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβουμε γιατί η πολιτική των μακροπεριφερειών ε, έχουν, ε, έχει επηρεάσει ε, τις δράσεις μου μέσα από τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο και αν δεν έχει αποδειχθεί, γιατί χάνουμε το χρόνο και το χρήμα μας για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Πώς πιτσιλ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα άκουσα με προσοχή. Εγώ εκπροσωπώ ψηφοφόρου τη Εθνική Δημοκρατίας και πιστεύουμε ότι ε, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διοχετεύονται σε διασυνοριακά προγράμματα και όχι σε εθνικά προγράμματα. Εφόσον μιλάμε για σειροδρομικές υποδομές, ε, θεωρώ ότι ε, ακόμη έχουμε πολλά να κάνουμε. Έπεσε το σιδηρό παραπέτασμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν συνδέονται με μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία επαρκώς, η Τσεχία με τη Γερμανία. Πώς γίνεται λοιπόν, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε την απαιτούμενη υποδομή. Χρειάζονται επενδύσεις. Εάν δεν επενδύσουμε στην διασυνοριακή συνεργασία, εάν δεν ε, καταφέρουμε ε, να αναβαθμίσουμε τις υποδομές, δεν πρέπει να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας και χρειάζονται επενδύσεις. 220 ε, εκατομμύρια έχουμε για την περιοχή του Δούναβη, μα δεν επαρκεί αυτό το ποσό. Δεν επαρκεί ούτε καν για τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών. Έχουμε κάνει μελέτες ε, για την ε, σύνδεση της ε, Πράγας με το Πίλσεν και την Ιρεμβέργη, ίσως και μέχρι το Μόναχο. 1,4 δις χρειάζονται δηλαδή πενταπλάσιο το ποσό σε σχέση με το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τον εξυγχρονισμό των υποδομών και γι' αυτό στο μέλλον θα πρέπει να συζητήσουμε για το αν τελικά είναι συμβολική η συνεισφορά μας μέσα από αυτά τα κονδύλια ή αν τελικά θα το πάρουμε στα σοβαρά και επενδύσουμε τελικά και για το τροχαίο υλικό. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει μόνο... Ε, ε, συγγνώμη για τους ποδηλατόδρομους, ε, σημαντικό και αυτό, αλλά δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε συνδροδρομική υποδομή. Εξαιρετικά τα προγράμματα, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα χρήματα. Δεν φτάνουν. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για αυτή την παρουσίαση. Μα ενδιαφέρει πολύ η μακροπεριφερειακή συνεργασία για να πάψουν οι ανισότητες και οι αποκλήσει μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Εδώ μιλάμε βεβαίω για τι δημόσιε υπηρεσίε του σιδηροδρόμους. Η διαλειτουργικότητα και καλή διασύνδεση της Ευρώπης ήταν ένα θαύμα της ε, αλληλεγγύης 10 δις ευρώ τα οποία προέκυψαν από τα διευθυντικά ταμεία. Ε, είναι πολύ περίπλοκο πλέον το δίκτυο, είναι περίπλοκη και η διαχείρισή του, όμως είμαι ιδιαίτερος ικανοποιημένη. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για διαδρόμους, νέους διαδρόμους και μάλιστα πολυτροπικούς όπως έχουν ονομαστεί, δηλαδή με διαφορετικούς τρόπους συγκοινωνίας. Ναι, ε, να θυμίσω ότι υπήρχαν οι νέοι διάδρομοι, οι πολυτροπικοί διάδρομοι, οι, οδικοί, ε, οι οδικές μεταφορές και οι πλωτή δρόμη. Η Ρουμανία βεβαίω δεν είχε υποβάλει εγκαίρω το εθνικό τη πρόγραμμα, τουλάχιστον επί τη προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα, πρόγραμμα αυτό υπευλήθη τελευταία στιγμή, αλλά τέλο πάντων υπευλήθη. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τις ανησυχίε κάποιων συναδέλφων όταν λένε ότι δεν υπάρχει αρκετό ποσοστό απορρόφηση των κομπηλίων, δεν υπάρχουν αρκετέ εγκαταστάσει, ότι δεν γίνονται αρκετέ επενδύσει στα τρένα υψηλή ταχύτητα. Να κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μιλάμε για τρένα που απευθύνονται στους τουρίστες ε, εκτός εάν κάποιοι δεν θέλουν να παραμείνει πλωτή οδό ο Δούναβης. Πάντω αυτά που μα έχει παρουσιάσει η κυρία Κρετσού είναι θαυμάσια από την άποψη τη ανάπτυξη και του τουρισμού. Να μην ξεχνάμε λοιπόν το τέταρτο, την τέταρτη δέσμη μέτρων για του σιδηροδρόμου και δημόσια υπηρεσία και να μην κοιτάζουμε μόνο τι δημόσιε κοινωνίε. Με συγχωρείτε, αλλά από τον κύριο Κόμπερν, ε, γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε, ωραία. Ευχαριστώ. Απλώς να πω ότι στην Βρετανία έχουμε κάνει τεράστια ασφάλματα γύρω στη δεκαετία του 50 όταν κλείσαμε πολλά από τα σιδηροδρομικά μα δίκτυα, τα μικρά επαρχηριακά δίκτυα, διότι θεωρούσαμε ότι δεν συμβατά με τι μελλοντικέ ανάγκε. Λέτε και συμφωνώ ότι το τρένα είναι το μέλλον. Όμω, έχουμε εξοδέψει ήδη πάρα, πολύ, πάρα πολλά στο SH2, το οποίο είναι ένα τρένο που πηγαίνει πολύ γρήγορα από την ε, Νότια Αγγλία στην Σκοτία. Αυτό που θα θέλαμε να έχουμε είναι ένα εύρωστο σιδηροδρομικό δίκτυο παρά να ξοδέψουμε μια περιουσία σε ένα πολύ ακριβό τρένο που δεν βοηθά τους μέσους ταξιδιώτες που χρειάζονται να μετακινούνται καθημερινά. Αστρονομικά ποσά και αυτό αφορά μόνο πολύ μεγαλόμιστους επιχειρηματίες και μέλη του δικού μας σώματος. Θα ήθελα λοιπόν χρήματα να δαπανώνται για τους μικρούς επαρχιακούς σιδηροδρόμους αντί να μεταφέρουμε το εμπόριο από τη μία περιοχή σε μία άλλη και όλα τα ενδιάμεσα να μένουν ξεκρέμαστα. Κοιτάξτε, ε, εγώ είμαι Ισπανίδα και πρέπει να αναγνωρίσω την επιτυχία που είχαν τα τρένα υψηλή ταχύτητα στην Μάλαγα, τη Σελβίνη, την Παρκελόνη. Έφεραν πολύ, πολύ περισσότερη εμπορική κίνηση. Η ισπανική εμπειρία ήταν αντίθετη από τη δική σα. Ε, είναι αλήθεια ότι, αν υπάρχει, ότι υπάρχει διαφορετική ε, πυκνότητα στον πληθυσμό, και στην ε, διανομή του στην επικράτεια της Ισπανίας. Δεν υπάρχει λοιπόν άμεση σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών, όμως σίγουρα χρειάζονται και δυνατότητες και δυναμικό για να μπορέσει κανείς να διαχειριστεί ένα καλό τρένο. Γιατί να μην υπάρχει ένα τέτοιο τρένο που να σας πάει απευθεία στη Σκωτία. Και ταυτόχρονα θα μπορούσε και να επικεντρωθεί στα μικρά επερχιακά δίκτυα, τα οποία είναι και αυτά πολύ σημαντικά. Οι πολίτες ε, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Ευχαριστούμε Γιάκοφτιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να τονίσω τρία σημεία, τρία προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, στις μακροπεριφέρειες, το να χρησιμοποιηθούν οι σιδηροδρομοί ως ένα εργαλείο θα απαιτήσει τεράστια δαπάνη κονδυλίων. Όμως, ε, το σημαντικότερο είναι να διασυνδέσουμε τις συνδρομικές με τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές. Έπειτα, ε, το άλλο που με απασχολεί είναι η απομόνωση των συνδρομικών δικτύων ε, και η παλαιότητά τους, λόγω χάρη γραμμή Αγκώνα Μπάρι ή όσα συμβαίνουν ε, στην Κροατία, Μπλότσεκ, Σεράγεβο, Ράντεν, Ζάγκρεπ και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν να τονίσω κάτι που μας ενδιαφέρει ως ιδιαίτερος για την Ίστρια. Οι σιδηρόδρομοι της Ίστριας μας διασυνδέουν μόνο με τη Σλοβενία. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει διασύνδεση με το συγχρονότερο δίκτυο των υπόλοιπων χωρών ή τουλάχιστον μια πρώτη συμφωνία με τις σλοβενικές αρχές. Ελπίζουμε να υπάρξει στήριξη μέσα αυτό το πακέτο γι' αυτό. Κύριε Γιάκοπτσιτς, μια μπλε κάρτα από την κυρία Σόλτες. Ναι, ναι, βεβαίως. Τον κύριο Σόλτες, τον κύριο Σόλτε. Και, και μετά άλλη μία κιόλα. Ο κύριος Σόλτες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάκοπτσίτς, αναφέρατε τη σύνδεση Κροατίας-Σλοβενίας όπως όλοι γνωρίζουμε μεταξύ του 1902 και 1935 υπήρχε η σύνδεση η Πορεζάνα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν ε, θεωρείτε πως υπάρχει περίπτωση να αναβιώσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Βεβαίως ε, το κροατικό κομμάτι των στυροδρόμων που συνδέεται με Σλοβενία μπορεί να λυθεί μέσω ενός τούνελ μέσω του όρους Ούτσκα αλλά αυτό κοστίζει και θα καθυστερήσει. Καλύτερο είναι να συμφωνήσουν οι δύο εταιρείε. Δεν βλέπω κάποιο λόγο. Γιατί δεν μπορεί όπως ήταν επί Ιουγκοσλαβίας ε, ε, Θα είχαν βρει. Αν μπορούσαν τότε να συμφωνήσουν, νομίζω μπορούν να το κάνουν και τώρα. Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν, το κομμάτι αυτό της γραμμής θα καταρρεύσει. Σας ευχαριστώ η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση. Συνάδελφε, είπατε πως είναι σημαντικό να συνδέσουμε αεροδρόμια και λιμάνια. Δηλαδή λείπει κάπου ο σιδηρόδρομος ή πρέπει να φτιάξουμε ένα σιδηρόδρομο αρκετά γρήγορο για να πετάμε λιγότερα, λιγότερο, όπως είπε. Όπως θα άρεσε και στον κύριο Κράμερ, άλλωστε. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να τονωθεί η, η διατροπικότητα στις μεταφορές. Μπορείτε στο βόρειο τμήμα της Αδριατικής ε, να πάτε εύκολα στο μπάρι, αλλά αν θέλετε από το μπάρι να πάτε στο Ριέκα, μετά ε, δεν μπορείτε να επιτύχετε ε, ταχύες μεταφορές. Δηλαδή θέλουμε ε, ναι, με σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά ταχύτερες. Επίτροπε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι διότι εξακολουθείτε να υποστηρίζετε την προσέγγιση αυτή με τις μακροπεριφέρειες. Τώρα συζητούμε την περιοχή του Δούναβη και της Αδριατικής. Δεν έχει σχέση μόνο με τη διασύνδεση των μακροπεριφερειών. Μάλλον την ε, απλή διασύνδεση δύο περιφερειών, αλλά ε, τις διασυνδέσεις στο εσωτερικό της μακροπεριφέρειας ε, για τη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων από τη βόρεια προς την Νότια Ευρώπη και αντίστροφα. Όμως δεν υπάρχουν εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές προς το παρόν. Δεν υπάρχουν διάδρομοι. Για τις εμπορευματικές λοιπόν μεταφορές ε, με σιδηρόδρομο θα πρέπει να σχεδιάσουμε νέους διαδρόμους και για την περίοδο 2014-2020 δεν καταλαβαίνουμε πού θα βρούμε τα κονδύλια από το ΣΕΦ, από το ε, χρηματοδοτικό μέσο για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν τέτοια προγράμματα. Ε, θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα και ανακατανομή των κονδυλίων για να υποστηρίξουμε και τις ε, υποδομές μεταφορές αλλά και την περιβαλλοντική πολιτική γιατί τους στόχους μας, είτε μιλάμε για τις μεταφορές είτε για το περιβάλλον, δεν πρόκειται να τους υλοποιήσουμε στα... στις προθεσμίες που έχουμε ορίσει. Για την ε, ανάπτυξη δρομικών ε, υποδομών θα πρέπει επίσης ε, να αυξήσουμε το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων και κυρίως να έχουμε διασυνοριακές υποδομές. Στην Κροατία έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Χάρη σε έναν διαγωνισμό κρατικών προμηθειών ναι, μπορείς να υλοποιηθεί ένα σχετικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να φροντίσουμε αυτές τις στρατηγικές να μας δώσουν χειροπιαστά αποτελέσματα και αυτό υπάρχει ένας τρόπος να γίνει, να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολιτών. Εάν κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή το δίκτυο του τι συμβαίνει στην διασύνδεση των ε, υποδομών των συγκοινωνιών, στην Αδριατική και τον Δούναβη, έχουμε ουσιαστικά μια τρύπα. Μια κενή τρύπα όπου δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Ε, καλό λοιπόν την κυρία Επίτροπο να διατρέξει όλη την ακτογραμμή της Αδριατικής με τρένο για να δει κατά πόσον ε, στους βασικούς άξονες αυτό το, αυτή η έλλειψη διασύνδεσης είναι τόσο εμφανής αρχή, η υπεύθυνη αρχή είχε τοποθετηθεί τον περασμένο Οκτώβριο για το θέμα αυτό και είχε εντοπίσει αυτή την απέτηση λέγοντας ότι σε όλη την αχοκοκαλιά της Αντρικής από την Αγκώνα μέχρι την Πεσκάρα και ως τον Μπάρι και τον Πρίντιζη πρέπει να ενισχυθεί η σιδηροδρομική διασύνδεση. Η Επίτροπος αποφε αποφασίζει να ε, επενδύσει στη γραμμή Τωρίνο Λιών, που είναι πολύ αμφιλεγόμενη, αντί να επενδύσει στην Νότια Ευρώπη, στην νότια πλευρά τη Αδριατική. Χρειάζονται περισσότερε επενδύσει ακριβώ για να καλυφθούν οι ελλείψει και η έλλειψη ισότητα που υπάρχει σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πρέπει να, να φανεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από όλα τα θεσμικά, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για όλε τι περιοχέ και του Νότου. Δείχνοντα ότι τη δική σα πλευρά υπάρχει υπεποίθηση ότι οι περιφέρειε του Νότου δεν θα πρέπει να χάσουν το ραντεβού με το μέλλον. Ε, οι πληρωμές έχουν αποφασιστεί και θα πρέπει να εκταμιευθούν μέχρι και προκειμένου η στρατηγική να επιτέχει τους στόχους της. Θα θέλαμε λοιπόν να φέρετε πλήρως εις πέρα στην ε, εκτέλεση των καθηκόντων σας. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε οι μηχανισμοί για τους οποίους μιλάμε σήμερα είναι σημαντικοί για τον Δούναβη και την Αδριατική. Σημαντικοί για τις συγκοινωνίες, ειδικά σιδηρόδρομο και δρόμους. Και βεβαίως ε, τα υφιστάμενα δίκτυα είναι κατακαιρματισμένα και περιορίζονται σε περιφέρειες ή και χώρες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να επεκταθούν οι συνδέσεις και να εξυγχρονιστεί το τροχαίο υλικό. Ε, το σύστημα των μακροπεριφερειών θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για αυτά. Και επίσης θα μπορούσαμε να δούμε και τι γίνεται και με τα μη καράτη μέλη. Ειδικά αν πρόκειται για χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη. Έτσι θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των μακροπεριφερειών Δούναβη και Αδριατικής και βεβαίως θα έχουμε και τις θετικές ε, επιπτώσεις και θα επιτύχουμε το λεγόμενο αποτέλεσμα αυτό του διαδρόμου. τα αποτελέσματα της συνέργειας ε, εντός ε, των μακροπεριφερειών ε, δεν τα έχουμε καταληφθεί πλήρως και εξακολουθούν να υπάρχουν στενοποί. Πρέπει λοιπόν να διασυνδέσουμε καλύτερα τις υποψήφιες χώρες και να δημιουργηθεί το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. Και εμείς θα βοηθήσουμε την Κομισιόν να βρει ρεαλιστικές λύσεις που θα συμφωνούν με όλα αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Φρουντσουλίκα. Ένα μισή λεπτό. Ο κύριος Φρουντσουλίκα. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ρουμανία για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου είναι πολύ καλός εταίρος, είναι εκτεταμένο το δίκτυο, μεγάλη ζήτηση για την κινητικότητα και λόγω του, της στρατηγικής της θέσης ε, στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών, ε, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στη Ρουμανία, υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις σε αυτό το τομέα και χρειάζονται ταχύτατα ε, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ε, φυσικά γίνεται ένα βήμα με το master plan 40 δις ε, θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα αυτό τον επόμενο χρόνο, κυρίως για την αναβάθμιση ε, σιδηροδρομικών γραμμών ε, μήκους 4.000 χιλιόμετρων. Όπως βλέπουμε στο Master Plan, η ε, BRD και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν ήδη επενδύσει από τις αρχές ε, του 90, όμως ε, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά και για τα αγαθά και για τη μεταφορά ανθρώπων. 2 και 3% και νομίζω ότι θα πρέπει να μειωθούν τα το λειτουργικό κόστος και να αυξηθεί η ε, λειτουργικότητα αυτού του δικτύου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακοπούν σιδηροδρομικές γραμμές. Ε, μην ξεχνούμε ότι όπως έχει κατάσταση στο σειροδρομικό δίκτυο της ε, Ρουμανίας θα απορροφηθούν όλα τα κονδύλια για την αναβάθμιση του δικτύου παρότι για το 2014 στο 2020 κατά μέσο όρο αυξάνεται κατά 2% ε, το κονδύλι για τις μεταφορές σε κάτι το παρελθόν όπου το ποσοστό ήταν 5% με την συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τον ίδιο αριθμό επιβατών με ένα μικρότερο δίκτυο από ό,τι φαίνεται κάποιες μελέτες ε, Κύριε Φραγκούλσα, από τον κύριο Κράμε δέχεστε μία μπλε κάρτα. Πολύ ωραία. Ναι, το ερώτημά μου βέβαια είναι το εάν το οδικό δίκτυο της Ρουμανίας είναι σε τόσο καλή κατάσταση που δεν σκέφτεστε να κλείσετε κάποιον δρόμο. Κάπου στην Ευρώπη κάποια στιγμή κλείνει κάποιος δρόμος γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για τη συντήρησή του. Το ερώτημά μου λοιπόν προβλέπετε στο master plan ένα 10-15% των δρόμων να κλείσουν ή κάνετε οικονομίες μόνο σιδηρόδρομους. Κύριε Φροντζουλίκα. Περιμένουμε τα κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα σιδηροδρομικά δίκτυα από ότι τους δρόμους, ε, κύριε Κράμερ. Ε, Ράντους, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Χαίρομαι που γράψαμε το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ε, οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ο φθηνότερος τρόπος μεταφοράς ε, και Κυρίως αυτή την περιοχή προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει διασύνδεση των πλωτών οδών με, τις, ε, με τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Και επίσης ε, ε, οι επενδύσεις που γίνονται σχετίζονται περισσότερο με τα οδικά και όχι τόσο με τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Η κυρία Κρέτσου είπε ότι τα TNT, τα διευρωπαϊκά, θα επεκταθούν στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα συνδεθούν καλύτερα με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά θα ενισχυθούν γενικότερα και τα ε, δίκτυα μεταφορών και έτσι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τις πλωτές οδούς περισσότερο. Σας ευχαριστούμε. Σνα... Στσάνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε το θέμα μας εδώ πέρα. Η περιοχή του Δούναβη είναι το 1 πέμπτο της έκτασης της Ένωσης και έχει το 1 πέμπτο του πληθυσμού. Η περιοχή αυτή ήταν πριν κομμάτι ενός άλλου μεγάλου σχεδίου ολοκλήρωσης πριν 100-150 χρόνια επίσης ο σιδηρόδρομος ήταν τότε σε άνοδο και τότε σιδηρόδρομος σήμαινε εξυγχρονισμός και αηφορία. Και σήμερα δεν διαφέρει πολύ το πράγμα. Ιστορικά γεγονότα οδήγησαν στον κατακαιρματιστεί αυτή η περιοχή. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει πάλι κάποια επανένωση θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε. Υπάρχουν επίσης ε, χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη και άλλες δύο χώρες που είναι εταίροι. Η Ουκρανία και, ο... και η Μολδαβία. Στην Ουκρανία υπάρχουν ακόμα και σήμερα κομμάτια του σιδηρόδρομου που δεν χρησιμοποιούνται αλλά μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όσον αφορά τα έργα τώρα, πιστεύω πως ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον να δούμε την διατροπικότητα και το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ. Μαμίκινς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από του ζωτικότερου τομεί ο σιδηρόδρομο στι δύο αυτέ μακροπεριφερειακέ στρατηγικέ, όπω ε, το σύστημα για την ε, ε, Ίστρια που ξεπερνά τα 230 εκατομμύρια ευρώ στην αξία του. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και τη συνοριακή συνεργασία και τη δημιουργία περισσότερων διακρατικών σιδηροδρομικών δικτύων που να είναι χρήσιμα για του πολίτε, αλλά να μπορούν να αξιοποιήσουν και τι υποδομέ. Το ίδιο ισχύει για την Αδριατική. Η διαχείριση της κυκλοφορίας ε, με την... Η καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας με περισσότερες επενδύσεις είναι σημαντικά. Ε, τα διευθυντικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια δυνατή πηγή χρηματοδότησης, αλλά για να ενισχυθούν αυτές οι δυνατότητες πρέπει να κοιτάξουμε και τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την επιβολή του νόμου και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, που και αυτά χρήζουν βελτίωσης. Αλλά χρειάζεται και η ανθρώπινη επικοινωνία και επαφή, διότι αυτή που είναι το μεγαλύτερο ε, Ευχαριστούμε. Ε, η διαδικασία κατστιάει τώρα. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γιασλοβιέτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική και τα δίκτυα TNT για την περιοχή του Δούναβη και της Αδριατικής. Συμφωνώ απολύτως με την ουσία της έκθεσης του συναδελφού που θέλει σχετικέ υποδομέ και καταστάσει να ε, αναπτυχθούν περαιτέρω σε αυτέ τι δύο περιφέρειε. Όμω θέλω να ρωτήσω την Επίτροπο τι επίπεδο προτεραιότητα ε, έχουν οι πλωτέ μεταφορέ στα πλαίσια αυτή τη στρατηγική, ιδίω για τον Δούναβη. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Αυτό το θέμα είναι μείζονος σημασίας, γιατί θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι ευτύχημα που μιλάμε για το θέμα αυτό τώρα. Η Ευρωπαϊκή Στατικική για τις Μεταφορές για την περιοχή του βούναβη και της Αδριατικής είναι ένα θέμα σοβαρότατο. Κυρία Επίτροπε, είπατε με σαφήνεια ότι σε κάποιες χώρες η ποιότητα των μεταφορών είναι αμφισβητήσιμη, όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας κλπ. Είπατε δεν ικανοποιείται και η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα απολύτως, αλλά είπατε ότι τρία πράγματα προέχουν για να βελτιωθεί η διαλογικότητα, η διαλειτουργικότητα μάλλον, οι επενδύσεις είναι ένα από αυτά. Μπορείτε να πείσετε τον κύριο Γιούνκερ, και αυτή είναι η ερώτησή μου, ότι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων χρειάζονται περισσότερα κονδύλια, περισσότερα προγράμματα, ώστε να ενισχυθούν αυτές οι περιοχές που έχουν μείνει πίσω. Δεν πιστεύω ότι η αγορά πρέπει να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα. Ε, οι επιχειρήσει πρέπει να να παρέμβουν και να καλύψουν το κόστος. Συμφωνώ λοιπόν με όσο είπε ο κ. Κράμερ και οι οδικέ μεταφορέ ε, προκαλούν ρήπανση μεν, αλλά και οδικά ατυχήματα, τροχαία και απώλεια ανθρωπίνων ζώων. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει τα κονδύλια να κατευθυνθούν στι περιοχέ που έχουν μείνει πίσω ω προ τι συνδρομικέ του υποδομέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία... Ε, κυρία Επιτροπέ, πήρα το τρένο από το Σαράγεβο μέχρι την δική σας πόλη και θα είχα κάνει 800 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόσο χρόνο θα μου χρειαζόταν, 48 ώρες. Είναι πολύ πιο απλό λοιπόν να έρθει κανείς ως εδώ, για να το πω έτσι, παρά να ταξιδέψει το Σαράγεβο και τη δική σας γενέτειρα. Ακόμη και αν είναι τέσσερις φορές μακρύτερη η διαδρομή. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει η ανενόχλητη ανάπτυξη του τουρισμού, της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών. Και γι' αυτό πραγματικά σας συγχαίρουμε για την πρόκληση που έχετε αναλάβει. Ελπίζω το στίχημα βέβαια αυτό να, να το κερδίσετε σύντομα με, ε, με καρπούς χειροπιαστούς, με χρηματοδότηση και με διαλειτουργικότητα που να γίνει πραγματικότητα στις ε, ε, συγκοινωνίες ώστε να σταματήσει να είναι μια, ένα σφουγγάρι με πολλές τρύπε το δίκτυο των μεταφορών στις μακροπεριφέρειες του Δουνάμι και της Η κυρία Κρετσού, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές για τις ε, παρεμβάσεις σας στην συζήτηση αυτή που μας δείχνει ξανά πόσο σημαντικές είναι οι συνδρομικές συνδέσεις. για τον Δούναβη και την εσωτερική αγορά. Να επισημάνω κάποια πράγματα όσον αφορά τις μακροπεριφέρειες. Ξέρετε πως δημιουργήθηκαν υπό τους όρους ότι δεν θα υπάρξουν νέα θεσμικά όργανα και νέες χρηματοδοτήσεις, οπότε ενώνουμε πόρους για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που δεν σταματάνε σε σύνορα και η Κομισιόν είναι απλά ένα συντονιστής. Τα προγράμματα, τα έργα τα κανονίζουν τα κράτη-μέλη και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ε, δεν μπορούν να φτιάξουν και να καθορίσουν αυτά τα έργα. Το θέμα λοιπόν είναι η συνεργασία των κρατών μελών με χώρες ε, εκτός ε, της Ένωσης και τώρα αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο να συνεργαστούμε με χώρες εκτός της Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινέ προκλήσεις όσον αφορά π.χ. την στρατηγική του Δούναβη. Μα μιλάμε εκεί πέρα για 40 χώρες. Ε, 14 χώρες, με συγχωρείτε. Εντός και εκτός ε, ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για υποδομές οι οποίες είτε δεν είναι ικανοποιητικές είτε δεν υπάρχουν ε, καν. Και συμφωνώ μαζί σας εγώ, ήμουν στο Σαράγεβο και για να πάω πίσω στο Βουκαρέστι έπρεπε να πάω μέσω Βιέννης ή Βρυξελών. Λοιπόν, οι υποδομές δεν υπάρχουν και όταν μιλάμε και για δύο συνοριακές διασυνδέσεις. Ε, δυστυχώς οι εθνικές αρχές δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Και το σχέδιο για τον δούνα ζητάει από τα κράτη-μέλη να κάνουν ακριβώς αυτό και θέλω να το επαναλάβω το μήνυμα αυτό. Δηλαδή να υπάρξει σύνδεση των υποδομών, ειδικά στις μεθοριακές περιοχές, ειδικά ο πληθυσμός ε, της υπαίθρου είναι υψηλότερο σε εμά από ό,τι στα άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τώρα τις θαλάσσιες μεταφορές και αυτό σχετίζεται με τη στρατηγική του Δουναβή. Και έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα εκτεταμένα. Και νομίζω πως πρέπει να τονίσουμε το ότι η συνδεσιμότητα και ειδικά η συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων είναι προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική του Δουναβή και του Ιωνίου και εγώ ήμουν ε, διαμεσολαβητής μεταξύ των Υπουργών Μεταφορών Βουλγαρίας και Ρουμανίας. είχαν τεράστια προβλήματα με τις ε, μεταφορές των Δούναβη γιατί είχε πέσει χαμηλά η στάθμη. Και προσπαθήσαμε να μεσολαβήσουμε, να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ των Υπουργών. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε Ε, είναι, είναι το πράγμα Δηλαδή ένα μέτρο πέφτει η στάθμη και από Ρουμανία μέχρι Γερμανία σταματάει η κυκλοφορία. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποια βήματα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά την περιφέρεια Αδριατικής ε, Ιωνίου περιλαμβάνει 8 χώρες. τέσσερα κράτη-μέλη και 4 μη κράτη-μέλη εγώ ευχαρίστω να πάω στο Ντουμπρόβνικ ε, όταν θα ξεκινήσει αυτή η στρατηγική. Κοιτάξτε, οι σιδηρόδρομοι τα πάνε καλύτερα, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωση, Υπάρχουν επίσης κάποια έργα στην περιοχή αυτή και βεβαίως χρειάζεται να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές των διευρωπαϊκών δικτύων. Και αδείχνουν πως η επιβατική κίνηση πέφτει όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα. πράγματα ακόμα. Χρειάζεται καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και ισχυρή πολιτική βούληση για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να επιτρέψουμε να ανταποκριθούν οι σιδηροδρόμοι στις απαιτήσει του πληθυσμού. Οπότε τώρα έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά την εργαλειοθήκη όπως λέμε για να προωθήσουμε τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες πιστεύουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σημειώσουμε πρόοδο για το περιβάλλον, τους πολίτες και την Ένωση στο σύνολό της. για λυπάμαι γιατί ο έφυγε. Ε, λέτε πως η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται για το νότο της Ευρώπης. Πληγώνουν αυτά που λέτε. Είχα πάει εγώ η ίδια δύο φορές εκεί πέρα. Α, η συνάδελφος είναι εδώ. Είχα πάει και στην Σικελία, Καλαβρία. Όταν είχα πάει στην Ιταλία ως Ευρωπαίος Επίτροπος ε, και ξεμπλοκάρισα τα έργα αυτά στην Νάπολη ξεκίνησε μια σιδηροδρομική σύνδεση που ελπίζουμε να λειτουργήσει εντός της ε, θητείας μας. Και συνδέθηκε η Ιταλία όχι μόνο από βορρά αλλά και από ανατολή προς Και τώρα ε, δεν θέλω να μπω συζήτηση αυτή για τη Ρουμανία απλά να σας πω ότι δεν επιλέγει η Κομισιόν τις προτεραιότητες Αυτά είναι στην εθνική στρατηγική. Είτε μιλάμε για τη Ρουμανία είτε όχι. Η Κομισιόν στηρίζει, οι υπηρεσίες Κομισιόν απλά στηρίζουν την διαδικασία. Ταυτόχρονα βεβαίως κάθε χώρα, κάθε κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να χαράξει τις προτεραιότητες της και εμείς δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ε, διαδικασίας η κυβέρνηση θα επιδείξει αρκετή ευελιξία για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τώρα λοιπόν.